Ε, και στο πολιτικό μέτωπο και στο μέτωπο της συνεργασίας ε, σε επαφή με τους ε, Νιγηριανούς ομολόγους μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε και πριν προχωρήσω παρακάτω μόλις πληροφορήθηκα ότι κάποιος ήθελε να θέσει διαδικαστικό θέμα επειδή δεν πήρε το λόγο στο Catch the Eye. Να πω ότι το Catch the Eye δεν είναι δικαίωμα, είναι μια δυνατότητα. Ο πρόεδρος αποφασίζει ποιος θα πάρει το λόγο ή όχι. Είχαμε πει ότι θα δώσουμε το λόγο σε δύο άτομα, έδωσα το λόγο σε πέντε. Λυπάμαι αλλά είσαστε μετά. Τώρα κλείνω τη συζήτηση και συνεχίζουμε με τις ψηφοφορίες. Πρέπει να ψηφίσουμε έξι σχέδια ψηφισμάτων για την κατάσταση του Τζιμπουτί. Υπάρχει μια, ένα κοινό ψήφισμα από πέντε πολιτικές ομάδες. Τροπολογία 1 της Γκουε. Ψηφίζουμε τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τώρα ψηφίζουμε το κοινό, ψηφίζουμε στο, σύνολο, του. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται Το επόμενο θέμα τώρα είναι έξι σχέδια ψηφισμάτων για την Ιγυρία. Αρχίζουμε με το κοινό ψήφισμα πέντε πολιτικών ομάδων. Τροπολογία 2. Ψηφίζουμε τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε καλύτερα. Έχω την εντύπωση εγκρίνεται, αλλά... Λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται όντως. Ψηφοφορία κατά τμήματα για την παράγραφο 18. Πρώτο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τμήμα 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. I put the vote to the motion for... Τώρα Ονομαστική ψηφοφορία για το σύνολο του ψηφίσματος. Παρακαλώ ψηφίστε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνετε. So, thank you very much for... Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.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 Κοιτάξτε, απλά ήθελα να κάνω μια παρατηρήση για τα πρακτικά τη χθεσινή συνεδρίαση που μα ε, διανεμήθηκαν στο σημείο 4 τη ημερήσια διάταξη, έγινε πολιτική συζήτηση επί των αποτελεσμάτων ε, τη Ιρλανδική Προεδρία και τη συμβιβασμού για τη Συμφωνία για το Πολιτέ Δημοσιονομικό Πλαίσιο αλλά τη στιγμή τη ψηφοφορία, δηλαδή στο σημείο 6 επί τη βάση του 169 παρενέβη ε, στο σημείο 6.2 αναφέρεται ένα ψήφισμα για τον απολογισμό της Ιρλανδικής Προεδρίας συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ψηφίσαμε ένα ψήφισμα και είναι ο τίτλος του ψηφίσματος για μια πολιτική συμφωνία για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020. Μήπως θα πρέπει να αλλάξουν λοιπόν τα πρακτικά και να μιλήσουμε μόνο για την πολιτική συμφωνία. Για τον απολογισμό της Ιρλανδικής Προεδρίας. Να είμαστε δηλαδή πιο σαφείς. Γιατί ήταν πολύ πιο συγκεκριμένος ο τίτλος του ψηφίσματος. Följegyezzük és tudomásul veszük, közvetítjük a megjegyzést. Ne, ναι, ne, ναι, πήραμε μήνυμα. Mr. Πρόεδρε, πολύ σύντομα να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ αυτή τη φορά γιατί επιτέλους είδα εδώ την κροατική σημαία. Χρόνια δούλευα για την υπόθεση αυτή. <coughs> Από τότε που ξε, που ήταν ακόμη εδώ ο Φον Χάμπσπουργκ το 1994. Θα ήθελα λοιπόν με αυτή την ευκαιρία να σε ευχαριστήσω εσάς και όλους τους συνεργάτες για τον τρόπο με τον οποίο ε, δούλεψαν τους τελευταίους 12 μήνες για μας όλους και να ευχηθώ καλές διακοπές σε όλους. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος. Πολύ καλά αυτά που είπατε, αλλά διαδικαστικά δεν ήτανε. Για τα πρακτικά τώρα θα υποβληθούν στην επόμενη σύνοδο δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα προωθήσουμε τα κείμενα που ψηφίστηκαν όπως δει και σας εύχομαι